θα αποσταλούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Υπάρχει θέμα διαδικαστικό. Παρακαλώ. Ε, thank you, President. I... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα στο πρώτο ψήφισμα για τη Ρωσία να καταγραφεί στα πρακτικά ότι υπερψήφισα το κείμενο. Αλλά δεν φάνηκε. Πάντως ε, το ότι στην πρώτη, στο πρώτο ψήφισμα υπερψήφισα το ε, σχετικό κείμενο. Ωραία.